Uh, Θα ήθελα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Δήλωση της Επιτροπής Εισαγωγή Συμβατών Συστημάτων για την ε, καταχώρηση κατοικιδίων Ζών στα κράτη-μέλη.